Okay. Mes chers collègues, j'ouvre notre séance. Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Επίσης, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ο Ζεράρ Ντεπρέ που είναι ο εισηγητής των άλλων τμήματων ε, του προϋπολογισμού του 2016 θα πρέπει να αποχωρήσει κατά τις 4 και 4 και 20. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα του δώσω την προτεραιότητα. Συμφωνείτε κυρία Γενική Εισηγητά. Ως προς τα πρακτικά της 3 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ να ζητήσω την έγκρισή σας διότι θα σας κοινοποιηθεί αργότερα το έγγραφο. Με την ε, ε, έγκριση, τη συμφωνία του Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντες θα δώσω το λόγο στο Ζεράρ Ντεπρέ. Άλλα τμήματα Κύριε Πρόεδρε, να πω και για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου δύο λόγια. Ναι. Ίσως αυτό είναι και το κύριο στοιχείο. Ωραία. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, Προσωπικά θα ήθελα να γίνουν ορισμένες προσαρμογές που θα αναφέρω. Ελήφθη μία απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρίου του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε παράρτημα αυτού του κειμένου της ε, Ολομέλειας, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά πριν από τις ε, θερινές διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Βασιζόμαστε σε αυτή την απόφαση δηλαδή. Δυστυχώς θα έχω ε, δυσκολίες με όλες τις τροπολογίες με βάση την πολιτική συμφωνία που έχει γίνει για αύξηση των πιστώσεων διότι είμαι υπόλογος της συμφωνίας που έγινε με το Προεδρείο. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που θα ήθελα να σας υποβάλω εντάχει. Καταρχήν είχαμε συμφωνήσει κατά τις διαπραγματεύσεις ε, με το Προεδρείο. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις γραμματείας, θα γίνει μία πρόταση τροποποίησης της ε, σύνταξης, γιατί δεν πρόκειται για αποζημίωση που αφορά τους βουλευτές που μπορούν να, την ε, να κάνουν χρήση και μπορούν να βάλουν τα χρήματα στην τσέπη τους. Διότι υπάρχουν ε, δημοσιογράφοι που ανέφεραν ότι πρόκειται για μία αποζημίωση των βουλευτών. Δεν, είναι κάτι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να γίνει λόγος για δαπάνες στη διατύπωση που σχετίζονται με το προσωπικό και τους παρόχους υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια των βοηθών των ε, βουλευτών θα αποφανθείτε εσείς ως προς αυτή τη διατύπωση για να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μια αποζημίωση που θα μπορούσαν να λάβουν οι βουλευτές. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου δεσμεύτηκε να δώσει τελική μορφή στις 3 Οκτωβρίου στην μεταρρύθμιση, στην αναθεώρηση του καθεστώτος των βοηθών των ε, βουλευτών. Αυτό είναι ευθύνη του προεδρίου και έχει δεσμευτεί να γίνει κατά την προσεχή συνάντηση της 3ης Οκτωβρίου. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του προεδρίου συμφώνησα επίσης για την εισαγωγή σε σχέση με το κείμενο που είχαμε εγκρίνει προγενέστερα ορισμένων τεχνικής φύσης τροπολογιών. Επειδή θα έχουμε πολλές πράσινες εβδομάδες, πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν, υπάρχουν και τα έξοδα ταξιδίου που θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 1.600.000 Άρα θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ε, αυξήσεις πιστώσεων, για παράδειγμα για τις στολές του, του, της υπηρεσίας ασφαλείας, για τους παιδικούς σταθμούς κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντιστάθμιση σε σχέση με τις ε, τακτικές δαπάνες. Συνοψίζοντας, η πρόταση που θα έκανα θα ήταν να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, ε, τη δέσμευση που λάβαμε με το Προεδρείο, με βάση την ποσοστή αναλογία που συμφωνήθηκε. Έχω υποβάλει μια τροπολογία για να ε, γίνει μια νέα διατύπωση σε σχέση με τη γραμμή των βοηθών και των ε, υπηρεσιών προς τους βουλευτές και θα υποβάλω και ορισμένε τροπολογίες όπως όρισε ο Γενικός Γραμματέας που είναι τεχνικής υφής και δεν θα έχουν επιπτώσεις σε σχέση με το γενικό προϋπολογισμό και το ύψος του. Όπως σας είπα, οι επικεφαλής ομάδων θα υποβάλουν τρεις τροπολογίες. Μία που σχετίζεται με την αύξηση των συμβασιούχων 43 για την ακρίβεια που θα διαθέτουν οι πολιτικές ομάδες. Επίσης, μία αύξηση της πυρκοδότησης των πολιτικών ομάδων της τάξης των 3.500.000 είτε για πρόσληψη είτε για ε, προαγωγές του προσωπικού και μία γραμμή για την τροποποίηση μίας θέσης Α10 σε AD14. Αυτά αφορούν τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι, νόμιζα ότι υπήρχαν ε, και άλλες λύσεις. Εγώ δεν δέχτηκα να υποβάλω αυτές τις τροπολογίες, γιατί εφόσον πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Δεν θα το κάνω εγώ. Φέρουν την ευθύνη οι πολιτικές ομάδες να υποβάλουν αυτές τις τροπολογίες και να τις προωθήσουν. Εγώ βασίζομαι στον, ε, και λαμβάνω θέση ως προς τον ε, προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εντάχει, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επίτηδες έλαβα υπόψη, σκόπιμα έλαβα υπόψη την ε, τροπολογία που υπέβαλε το ίδιο το θεσμικό όργανο, διότι Ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την αύξηση του αριθμού των δικαστών που υποστήριξε η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο σε σχέση με τη Γραμματεία γιατί ε, δεν ξέρουμε με βάση ε, τα δεδομένα του αριθμού των δικαστών δεν θα υπάρχουν στενοποί που δημιουργούνται όταν μειωθεί το προσωπικό υποστήριξης. Αυτό ζητήθηκε από το ίδιο το θεσμικό όργανο. Και ε, η γραμμή είναι λίγο υψηλότερη από αυτή που είχε εισαγάγει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο τώρα, δέχτηκα την πρόταση του ίδιου του θεσμικού οργάνου προσθέτοντας 100.000 ευρώ για ασφάλιση για μια ασφάλεια με στα πλαίσια του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που είχε διαβιβαστεί από την Κομισιόν μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προτάσεων. Πρόκειται για τα, τις 100.000 επιπροσθέτως που ζήτησε η Κομισιόν. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόωθησε αυτή τη θέση σε σχέση με την ΕΟΚΕ επαναλαμβάνω την πρόταση του ίδιου του θεσμικού οργάνου, τη δέχομαι, που δέχτηκε και η Επιτροπή. Μιλάμε για 36 θέσεις, ένα σχέδιο που προβλέπει 30 θέσεις, όπου μπορεί να γίνουν και μεταφορές όπως είχε συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και η ΕΟΚΕ. Σε σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών ήρθα σε επαφή με τις υπηρεσίες και διαπραγματευτήκαμε. Πρόκειται για μια θέση παρόμοια με αυτή της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά λίγο κατώτερο είναι το, το πλαίσιο, γιατί μειώσαμε ορισμένες θέσεις εργασίας και θεωρήσαμε ότι μειώθηκαν οι θέσεις ε, καταναλογίαν των αναγκών του θεσμικού οργάνου για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ε, δέχτηκα τις προτάσεις της Επιτροπής ως προς την αποκατάσταση του σχεδίου του προϋπολογισμού το ίδιο και για τον Ευρωπαίο Επόπτη των Προσωπικών Δεδομένων. Έχω ένα πρόβλημα όμως με την ΕΙΕΔ γιατί η Ε.Ε. όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ε, είναι μια δικέφαλη αρχή. Διότι επικεφαλής είναι η Αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπος και του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Άρα η ευθύνη και η λογοδοσία ε, αφορά έναν επιμερισμό αρμοδιοτήτων, επιτροπής και συμβουλίου. Άρα οι προτάσεις ε, διαφέρουν μεταξύ τους. Η Επιτροπή δέχτηκε τις ε, προτάσεις της ΕΙΕΒ κάθε αυτής και αυτό εξηγείται γιατί η κυρία Μογκερίνη είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα ήταν πολύ δύσκολο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ε, ε, δεχτεί τις θέσεις της Αντιπρόεδρου. Το Συμβούλιο ήταν ε, ήρτηρο και δέχτηκε μια αύξηση 3,79% αφού εξετάσαμε τις θέσεις του προϋπολογισμού και τα ποσά που πρότεινε η Επιτροπή και τις μειώσεις του Συμβουλίου βρήκα μια χρυσή τομή δηλαδή το μέσο όρο των αυξήσεων που προβλέπει η Επιτροπή και των ποσών που δέχεται το Συμβούλιο, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι πήραμε θέση υπέρ του Συμβουλίου και ή ότι δεχτήκαμε απολύτως τη θέση της Επιτροπής. Αυτό θα το δούμε στις συζητήσεις σε κάθε γραμμή του προϋπολογισμού. γιατί αυτή ήταν και η πιο λογική οδός. Αυτά μπορώ να πω, Πρόεδρε, σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων έχουμε λάβει πολλές ε, τροπολογίες από, από κάποια νέα ομάδα όπου ζητήθηκαν 43 θέσεις βοηθών αλλά έγινε πρόταση για μια συνολική μείωση 100 εκατομμυρίων ευρώ και από άλλες πολιτικές ομάδες έλαβα τροπολογίες τις οποίες θα συζητήσουμε πριν ψηφίσουμε, όπως ισχύει για κάθε τροπολογία ξεχωριστά. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις επικρίσεις αλλά και τις φιλοφρονήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αναφίβολα θα καταφέρουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε και στις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και στους ε, προέδρους των ομάδων, γιατί πρέπει να υπάρξει και μια αιτιολόγηση. Γιατί σε ό,τι αφορά ε, επιπλέον πιστώσεις υπάρχουν πολύ ισχυροί περιορισμοί και το κύρος μας θα εξαρτηθεί και από την εξέταση των ε, πιστώσεων που έχουν προταθεί. Ποιο θέλει να πάρει τον λόγο τώρα επί του ζητήματο αυτού. Κανείς δεν ζητά το λόγο. Σας έπεισα, λέει ο κύριος Δεπχέ. Είστε ιδιαίτερα πιστικός, κύριε Σιγητά. Και καθώς δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, ας ε, κλείσουμε αυτό το ζήτημα και να δώσουμε το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, Γενικό Εισηγητή, για να μας παρουσιάσει τη δική του θέση, γιατί ξέρουμε ότι σήμερα το ΕΚΟΦΗΝ ε, επιβεβαίωσε τη θέση της Κορεπέρ και υποθέτω ότι και οι επικρίσεις που διατύπωσε ο Χωσέ Μανουέλ πριν από δύο εβδομάδες σίγουρα θα τις επιβεβαιώσει και αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Οι επικρίσεις προς το Συμβούλιο ισχύουν, αλλά σήμερα θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες, τους ε, συναδέλφους και την εργασία τους μέσα στα πλαίσια των τροπολογιών. Να συγχαρώ την εξαιρετική μας ε, γραμματεία καθώς και τους ε, πολιτικούς ε, συμβούλους, γυναίκες είναι ε, σε αυτή την περίπτωση, γιατί χτες την Κυριακή ολοκλήρωσαν την εργασία από τις 10 το πρωί, αναλύσαμε όλες τις τροπολογίες και γι' αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.824 τροπολογίες. 1.824. ...532 από τις επιτροπές, 647 ε, ε, από τις ε, πολιτικές ομάδες, στη στήλη 1 στήλη 2 και 248 στη στήλη 4, 289 στην στήλη 5. Εάν ε, προσθέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε σχέση με το ε, σχέδιο του προπολογισμού, θα είχαμε αύξηση 50 δις ευρώ συνολικά, αν ελαμβάνονται υπόψη όλες. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες όλες, μικρές και μεγάλες. Αλλά αυτό δεν θα ήταν ε, ρεαλιστικό. Έχουμε ένα μικρό προϋπολογισμό που αντικατοπτρίζει το 1% των εθνικών ΑΕΠ. Θα σας κάνω μία ανάλυση των δεδομένων έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία συνένεση. Δεν νομίζω ότι θα είναι δύσκολη η συνένεση. Έχουμε μία σαφή στρατηγική και μία εντολή η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο από την Ολομέλεια και γι' αυτό οι πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές δέχτηκαν αυτή την εντολή, αυτή την ισχυρή εντολή. Αναλάβαμε ένα συμβιβασμό μέσα στα πλαίσια της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας μέσα στα πλαίσια και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στα πλαίσια των δαπανών. Όταν παρουσιάσουμε τις γενικές γραμμές του προπολογισμού, είπαμε ότι τα θέματα των ε, μεταναστών και των προσφύγων είναι ύψης της σημασίας και τώρα παραμένει στο επίκεντρό μας. Και αυτό φαίνεται και από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Δηλαδή οι πολιτικές ομάδες και οι συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα και το κεφάλαιο 3 θέλουν να το δουν στο σύνολό του, διότι υπάρχει το μέσο της εποπτείας, το μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας στη Μεσόγειο, το μέσων ε, για την προσχώρηση, η πρώτης ε, προσχώρηση. και άρα έχουμε όλα τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε οι οργανισμοί να ασχοληθούν με το θέμα. Τα πιλωτικά σχέδια που σχετίζονται με αυτή τη θεματική θα πρέπει να ειδωθούν στο σύνολό τους και ελπίζω και το ε, Συμβούλιο να έχει την ίδια ευαισθησία και να αναγνωρίζει πλήρως το θέμα και να δεχτεί και αυτή τη στοχοθέτηση, αυτό το πακέτο, έτσι ώστε να έχουμε επαρκής ποσά για να ελαχιστοποιήσουμε το δράμα που ζούμε στη Μεσόγειο. Βεβαίως θέλουμε ένα φιλόδοξο προπολογισμό, αλλά και ρεαλιστικό. Γι' αυτό για κάθε τροπολογία θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση, αντικειμενική αιτιολόγηση, μέσα στα πλαίσια του καθολικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα πρέπει να προβλέπονται επιμέρους ε, earmarkings. Όπως ε, ελέγχθη, θα χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα ευελιξίας και κάθε ευελιξία στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητές μας που θα πρέπει να είναι προτεραιότητες και του Συμβουλίου. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε ανακεφάλαιο, μέσα στα πλαίσια της τήρησης των συμβιβασμών, θα ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από τις ε, επιτροπές και τις ε, πολιτικές ομάδες, διότι δέχτηκαν τον, ε, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη και το μέσον Ευρώπη 2020. Και στο 1α, στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 και του συνδέοντας την Ευρώπη, προσπαθούν να λάβουν υπόψη και τα δεδομένα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Όπως προβλέπεται συνεργατικά από τα τρία θεσμικά όργανα. Για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτών των δύο προγραμμάτων, δηλαδή Ευρώπη 2020 και του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτά τα δύο μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικά για θέματα ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πρόθεση της απασχόλησης. Άρα, το σχέδιο Juncker και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αφορούν μία πρόταση μέσα στα πλαίσια του συμβιβασμού στον οποίο έφτασαν τα τρία θεσμικά όργανα και προσυπέγραψαν, που θα πρέπει να δούμε ξεχωριστά όταν δούμε τις επιμέρους προτάσεις του προϋπολογισμού. Ε, ορίζοντας 2020 έχει ενισχυθεί κατά 170 εκατομμύρια ευρώ και το συνδέοντας Ευρώπη έχει ενισχυθεί και κατά 120 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν και ε, προγράμματα όπως το Εράσμος, το Κόσμο και άλλα που έχουν ενισχυθεί, όπως ακριβώς ε, ζητήθηκε. Στο 1β, στην κεφαλίδα 1β, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόθεση για πρωτοβουλίες υπέρ των νέων. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνεχιστούν και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για έξι δις που προβλέπονται αρχικά έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία να συνεχιστεί. Επίσης, Υπάρχουν προτάσεις ε, τροπολογιών για να φτάσουμε στην τήρηση και του σχεδίου πληρωμών, δηλαδή να μην θίξουμε τα προγράμματα τα οποία τώρα τρέχουν. Και γι' αυτό οι πολιτικές ομάδες ε, μίλησαν για ένα δις για την Ελλάδα, για προκαταβολή, έτσι ώστε αυτό να φανεί σε, αυτό το, σε αυτή την κεφαλίδα. Και υπάρχουν και οι κατάλληλες τροπολογίες και για την ε, πρωτοβουλία υπέρ των νέων ε, υπάρχει ένας πολύ καλός ε, δείκτης εκτέλεσης και υπάρχει σωρία τροπολογιών. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις κεφαλίδες όπου υπάρχει ένας καλός δείκτης εκτέλεσης και όχι εκεί όπου δεν υπάρχει σωστή απορρόφηση. Στο, στον τομέα 2 επίσης στην, κεφαλία, στην κεφαλίδα 2 υπάρχει ένα περιθώριο 88 ε, δις Ευρώπη και, στο... και αυτό ισχύει και στην 1α. Ε, στην 2 πρόκειται για 152 δις. Όπως σας είπα, στο, στην κεφαλίδα 3 θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την έκτακτη ανάγκη που απορρέει από την κρίση των προσφύγων. Αυτός ο τομέας θα πρέπει να επανειδωθεί μαζί με το κεφάλαιο 4 στα πλαίσια των οργανισμών των πιλωτικών και των πιλωτικών σχεδίων. Οι προτάσεις τροπολογιών έχουν υποβληθεί από τις Επιτροπές. 89 είναι αυτές οι προτάσεις και οι πολιτικές ομάδες υπέβαλαν 109 προτάσεις τροπολογίας για τους οργανισμούς και για τα ταμεία. Στην κεφαλίδα 4 θα πρέπει να υπάρξει ε, μία σύνδεση μεταξύ των τεσσάρων προγενέστερων κεφαλίδων και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Ε, προβλέπεται μία αύξηση από τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη σύγκληση των πολιτικών ομάδων και η πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με το δεύτερο σχέδιο βοήθειας έχει ήδη εγκριθεί μέσα στα πλαίσια των ε, τροπολογιών. Μιλάμε για 172 εκατομμύρια και 390 εκατομμύρια αντίστοιχα για υποχρεώσεις και πληρωμές. Και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση προς την Επιτροπή με την ευκαιρία, εάν μπορεί να μας επιβεβαιώσει, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ότι για αυτή τη δεύτερη πρόταση, τα 180 εκατομμύρια ευρώ και 390 ε, για πληρωμές είναι ένα τελικό ποσό και κατά πόσο θα υπάρχει διορθωτική επιστολή, για να ξέρουμε δηλαδή κατά πόσο αυτά τα ποσά είναι τα τελικά ή θα αλλάξουν από την διορθωτική επιστολή. Για το πρώτο πακέτο, για τους 40.000 ε, πρόσφυγες, θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο προβλέπεται μία αύξηση και κατά πόσο θα ακολουθήσουμε την ίδια συλλογιστική που ισχύει στο δεύτερο πακέτο. Δηλαδή, τα χρήματα που θα δοθούν στις ε, χώρες υποδοχής, δηλαδή την Ιταλία, Ελλάδα. Δηλαδή, 500 ευρώ πρόσφυγα συμπληρωματικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πώς θα υπάρξει διορθωτική επιστολή και εδώ. Σε σχέση με το κεφάλαιο ή τομέα 3, στο 4 θα υπάρξει μία μικρή αύξηση. Στο κεφάλαιο 4, επειδή υπάρχει σύγκληση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αυτή τη βδομάδα θα φτάσουμε σε μία συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες για αυτό το τελικό στόχο. Θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ως προς τη δημοσιονομική μας στρατηγική, αλλά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και ως προς την ε, κρίση των προσφύγων. Ως προς τον τομέα 5 ακολουθούμε τη γενική μας ε, στρατηγική, όπως φαίνεται και από τις τροπολογίες, δηλαδή να γίνει μια αποκατάσταση του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής και άρα και στον τομέα η κεφαλίδα 5 ισχύει αυτός ο γενικός κανόνας. Ως προς τα πιλωτικά σχέδια τώρα, Είχαμε μεγάλη συμμετοχή και από τους συναδέλφους και από τις επιτροπές. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Έχουμε 218 πιλωτικά σχέδια. Τα ποσά είναι πολύ μικρά και έχουμε πολύ λίγα περιθώρια. Θα καταβάλουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια έτσι ώστε σε κάθε τομέα να έχουμε περιθώρια για αυτά τα πιλωτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 310 εκατομμύρια ευρώ σε, υποχρεώσεις. Και χωρίς να μπούμε στο θέμα των οργανισμών, γιατί υπάρχει ένας μόνιμος εισηγητής για τους οργανισμούς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλες τις πολιτικές ομάδες, διότι ε, ενίσχυσαν και υποστήριξαν τις εργασίες μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εξαιρετική εργασία της Γραμματείας, γιατί χωρίς εκείνη δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η εργασία του εισηγητή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Merci, monsieur le rapporteur Ευχαριστώ κύριε Γενική Εισηγητά και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ευχαρώ για την αφοσίωσή σας, τη διαθεσιμότητά σας ακόμα και όλες αυτές τις στιγμές ε, που ζήσατε μέσα στο πλαίσιο βεβαίως και μιας ε, ομάδας ε, με μεγάλη προγνωμοσύνη και όλοι σας πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ο Χασέ Μονέλ μας ε, ενημέρωσε σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επί του προπολογισμού. Μας είπε ότι θα πούμε σε μια πολύ δύσκολη φάση γιατί θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί η Ευρώπη διέρχεται μια πραγματικά μεγάλη κρίση, η ελληνική κρίση αρχικά, που μένει ακόμα να αποδειχθεί ότι οι δεσμεύσεις που έχουν ε, γίνει θα τηρηθούν. Και από αυτή την πλευρά μπορούν να υπάρξουν και ερωτήματα. Και μετά έχουμε και αυτή την ε, πραγματική μαζική φυγή και έξοδο ε, που θέτει στο πεδίο των διαπραγματεύσεων ε, όλη μας την πολιτική, στρατιωτική οντότητα, την αλληλεγγύη την Ευρώπη στο σύνολό τη, αλλά και τα κράτη-μέλη πιο συγκεκριμένα που ασκούν τα δικαιώματά του ε, ε, σε ένα πλαίσιο γενικότερης ε, ταραχής και χάους. Επομένω, αυτό ο προπολογισμό με πολύ σημαντικού περιορισμού, αυτό ο προπολογισμό με πολύ σημαντικού περιορισμού, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στα μέλη. Ο κύριος Φεζά που ήταν και στην Επιτροπή, εφόσον ε, υπήρξε το ερώτημα για την ιδιορθωτική επιστολή από τον κύριο Φερνάντε, θα θέλατε να μα ενημερώσετε, κύριε Φεζά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, ο κύριος Φερνάντες έθεσε λοιπόν δύο ερωτήματα. Κατά πόσο οι πιστώσεις ε, πληρωμών που θα είναι απαραίτητε για αυτό το δεύτερο πακέτο για τη μεταναστευτική ροή και την επανεγκατάσταση των προσφύγων ε, θα αποτελέσει αντικείμενο της θρησκευτικής επιστολής. Η απάντηση είναι ναι. Θα συμπεριληφθεί στη θρησκευτική επιστολή λοιπόν αυτό το θέμα που θα υποβάλουμε στα μέσα Οκτωβρίου μαζί και με τα πιο παραδοσιακά στοιχεία της θρησκευτικής επιστολή Περνώ τώρα στο δεύτερο ερώτημα του εισηγητή σε ό,τι αφορά τη διαφορά μεταξύ των δύο πακέτων. Πάντα σε σχέση με τη μετανάστευση. Το πακέτο του Μαΐου και το πακέτο που μόλις ε, ανακοινώθηκε. Εδώ υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία διαφορετική. Στο πακέτο του Μαΐου έχουμε προχωρήσει πολύ. Και ανεξάρτητα από την, ε, το τελικό αποτέλεσμα θα υπάρξει προσαρμογή του αντικτύπου στον προπολογισμό. Γιατί, όπως είπε και ο συγκητής, στα μέτρα που προτάθηκα τον Μάιο δεν υπήρχαν κάποια στοιχεία που έχουμε σε αυτό το νέο πακέτο μέτρων. για να πάμε πέρα από τα όσα είχαμε φανταστεί πριν από μερικούς μήνες. Με η διδακτική επιστολή ε, θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα τις ε, προοπτικές του υπολογισμού με βάση και τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί μέχρι τότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις βάθος του. Τα όσα είπε για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής γεωργίας που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε απασχόληση έχουν ουσιώδη σημασία, καθώς επίσης και για τους γνωστούς λόγους και τα όσα θα πρέπει να προσαρμόσουμε, να διορθώσουμε όσον αφορά βέβαια τις επιπτώσεις του πακέτου Juncker. Τώρα, έχετε δίκιο βέβαια λέγοντας ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα μετακίνηση πληθυσμών όταν τους επόμενους έξι μήνες, ή μάλλον αν τους, τους επόμενους έξι μήνες δεν έχουμε καμιά καλύτερη ιδέα από αυτές που είχαμε το προηγούμενο εξάμεινο, τότε θα πρόκειται για πραγματική ανθρωπιστική καταστροφή. Πρόκειται για μια κίνηση πληθυσμών που θα μας απασχολήσει για δεκαετίες. Και θα αποδειχτεί ότι οι περίφημες αξίες που θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε θα, δεν θα έχουν καμιά απολύτως αξία και θα επαληθευτεί αυτό που έλεγε κάποιος ότι υπνοβατώντας πήγαμε στην καταστροφή. Δεν κατανοώ λοιπόν πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει τόσο γαλήνια όταν έγινε ένα σοβαρό βήμα την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή πρότεινε ένα πακέτο μέτρων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλές από τις πτυχές αυτών των μεγάλων θεμάτων και σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική αυτή θεομηνία και μια συνολική στήριξη. Πρόκειται ωστόσο για ένα πρώτο πακέτο μέτρων που θα αποδειχθεί στο τέλος ότι δεν είναι επαρκές. Ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών χθε σε μια συνέντευξή του online είπε ότι από μια στιγμή και μετά αντιμετωπίζουν υπερβολικό βάρος οι χώρες που αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Και πολύ σύντομα και οι χώρες που δέχονται τώρα τους μεγάλους αριθμούς των προσφύγων, πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσουν και αυτές τα όρια τους. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ήδη ότι αυτά τα πρώτα hot spot, αν θέλουμε να λειτουργούν, αυτό θα γίνει μοναχά εάν γίνει και η περαιτέρω κατανομή και έχει συμφωνηθεί δηλαδή η παραπέρα κατανομή των προσφύγων και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αν δεν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τους αριθμούς πρώτα των 40.000, δεύτερα των 160.000 που ίσως και να μην τα καταφέρουμε το ερώτημα που θα τεθεί είναι και τι θα κάνουμε με τα υπόλοιπα που μας έρχονται. Πρόκειται για πραγματική, θα είναι πραγματική αποκάλυψη με την έννοια της αποκάλυψης. να. Πρόκειται για λοιπόν μια πρώτη κατανομή και εκεί προβλέπουν περίπου 98 εκατομμύρια για το εργαλείο ευελιξίας και φαίνεται πως το ΕΚΟΦΗΝ επιβεβαιώνει τα νούμερα αυτά. Και λένε τώρα για το τετραπλάσιο, άρα δηλαδή περίπου 400 εκατομμύρια. Γιατί πράγμα μιλούμε. Όταν θα ψηφίσουμε αρχές Οκτωβρίου τον προϋπολογισμό και θα έρθετε μετά από 10 μέρες και θα μας υποβάλλετε διορθωτική επιστολή που θα περιλάβετε εκεί και τι ιδιαίτερε ενισχύσει, τι ειδικέ ενισχύσει μάλλον για τη γεωργία. Νομίζω δεν ανταποκρίνεστε στην πραγματικότητα έτσι. Και να δούμε και τα νούμερα του Συμβουλίου που σε πολλά σημεία κάνει παραπάνω από ό,τι για το 2015, όμω, ορισμένα από τα νούμερα του που βάζει και στο 2015 είναι προχθεσινά. Ήδη βλέπουμε ότι ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στον Λίβανο δεν διαθέτει παραπάνω από το 1 τρίτο των κονδυλίων που είχε στην αρχή. Όταν βλέπω λοιπόν τι κάνουμε με τα διάφορα κονδύλια για την πολιτική γειτονία, προενταξιακά κλπ. Δηλαδή τι σκέπτεται να κάνει με αυτά τα πράγματα το Συμβούλιο. δεν ξέρω καν αν πρόκειται για σκάνδαλο ή πρέπει να χρησιμοποιήσω καμιά βαρύτερη λέξη. Αν λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες δεν καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στα στρατόπεδα προσφύγων, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγιεινής, προμήθειας των απαραίτητων, πάλι οι άνθρωποι θα ξεχωριστούν να φύγουν από αυτά τα στρατόπεδα προσφύγων. Και δεν θα μπαίνει πια μόνο το θέμα της Ουγγαρίας, υπάρχει και η Σλοβενία, η Κροατία, και θα αρχίσουν να πηγαίνουν πλέον μέσα από Ουκρανία και ε, Ρωσία για να φτάσουν στα βόρεια σύνορα της Ευρώπης και να μπουν από εκεί. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπους τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά εντατικότερα με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και πιστεύω ότι η Κομισιόν για το σύνολο των, των κονδυλίων στις κατηγορίες 3 και 4 που λέει ο εισηγητής να φτιάξει ένα κατάλογο, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε με τα διαθέσιμα κονδύλια. Πού θα πάνε τα κονδύλια αυτά, ποιο είναι δικαιούχο, ποιε δυνατότητε θα έχουμε, ποιε δυνατότητε έχουμε για να βοηθήσουμε στα στρατόπεδα προσφύγων. τι γίνεται με τα κονδύλια για να αναπτύξουμε τα λεγόμενα hot spot με άλλα πράγματα όπως ταμεία προσφύγων. Ποιοι θα είναι δικαιούχοι, ποιοι και πώς θα λάβουν τα χρήματα. Για να λάβουμε μία ανάλυση για το ποια πράγματα θα είναι αναγκαία πλέον το 2016 και από πού θα βρεθούν οι πόροι τους οποίους θα χρειαστούμε. Και αν υπάρχει προοπτική να τους βρούμε ή όχι. και το κείμενο της Κόμισιον της και δίνει απαντήσεις και που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο την προηγούμενη εβδομάδα και για αυτά τα trust fund που λέει σωστό το βρίσκω το κείμενο αυτό με συνεισφορές από τις χώρες, μάλι, ε, χώρες μέλη. Είναι ανοιχτό όμως εκεί. Ωραία ακούγεται αυτό το 8,1 δισεκατομμύρια. Το εάν όμω θα μπορέσουν να γίνουν οι μεταφορέ κονδυλίων από άλλε γραμμέ του προπολογισμού, αν πραγματικά θα γίνουν ή αν θα παραμείνουν σε αυτό το γνωστό πέρα δόθε μέσα στον προπολογισμό, για αυτό το πράγμα εγώ θέλω να δώσω συγκεκριμένου αριθμού, συγκεκριμένα νούμερα, για να μπορώ και να τα αιτιολογήσω. Γι' αυτό νομίζω πρέπει ίσως να συνοψίσουμε το ερώτημα αυτό, να το δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τους εξηγήσουμε ότι θέλουμε μια ξεκάθαρη ανάλυση τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα αυτά, με τα κονδύλια αυτά, με τους πόρους αυτούς, να δούμε εάν μπορούμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Διότι αλλιώ δεν μπορούμε. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μα δεν είναι μόνο θέμα πιστώσεων, είναι και θέμα γενικότερης οργάνωσης και συντονισμού. Δεν αρκεί να εγγράψει κανείς πιστώσεις, κονδύλια, πρέπει να σκεφτεί και τι θα κάνει για να ελέγξει αυτά τα, κύμα, τα, τα κύματα μετανάστευσης. 28 χώρες μέλη σημαίνει 28 διαφορετικές ρυθμίσεις οι πρόσφυγες. Έχουν, είναι και διαφορετική. Η ζήτηση για ορισμένε χώρε μέλη είναι λίγες μέρες, για άλλες είναι το λιγότερο σε βάση έτους σε ορισμένε χώρε θα λάβουν αποζημιώσει πολύ υψηλότερε από τις άλλε. Σε ορισμένε χώρε μέλη θα μπορέσουν να βρουν δουλειά αμέσω. Σε άλλε χώρε μέλη ίσω χρειαστεί να περιμένουν ένα χρόνο. Άρα στη βάση αυτών θα επιλέξουν και οι πρόσφυγε. Μια χώρα ή μια άλλη. Το να βάλει κανεί ποσοστώσει, ωραία, αλλά πάνω σε ποια βάση θα του προσανατολίσουμε. Υπάρχουν πολλά κενά και δεν έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρώπη έχει κατανοήσει ακόμα. Πήγα στην Ελλάδα, στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα οργανώνουν τη μεταφορά από τα νησιά, από την Κό και τη Λέσβο, κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη για να πάνε μετά στη Μακεδονία. Ναι, μπορείτε να ξεχάσετε επομένω τι συμφωνίε του Δουβλίνου. Σε όλη αυτή την περίοδο οι Ευρωπαίοι ασκούν οξύτατη κριτική στην Ευρώπη και αναρωτιόνται έχει τη δυνατότητα να δείξει ότι είναι μια πραγματική δύναμη η Ευρώπη κύριε Τελανό. Είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεση του προπολογισμού 2016 γιατί πέφτει πάνω σε διάφορες κρίσεις. Κρίση των προσφύγων που περιέγραψε καλά ο συνάδελφος Μπέκε και συμφωνώ εγώ με την προσέγγιση του. Υπάρχει η κρίση της ανεργίας των νέων, η κρίση του ελληνικού χρέους και βέβαια η κρίση στη Γεωργία που είναι και αυτή πολύ σχηδής και που συνδέεται σήμερα και με το ρωσικό εμπάργο αλλά και με άλλα με ε, ζωνόσους στην εκλογική μου περιφέρεια εμφανίζεται ε, ο αυτόδης πειρατός στα ζώα. Ε, σημαίνει πάρα πολλές δυσχέρειες αυτές στο μέλλον. Δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν εμπορικές κινήσεις ε, εκτός των ζωνών. Θα χρειαστεί να εμβολιαστούν οι αγέλες των βοηδών, κάτι το οποίο είναι δαπανηρότατο, θα κοστίσει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε λοιπόν εν μέση κρίση σε όλα τα επίπεδα και πρέπει πραγματικά να γίνει τεράστια προσπάθεια για να μπουν αυτά τα πράγματα μέσα στον προϋπορισμό και συγχαίρω τον φίλο Φερνάντες. Χρειάζεται να ασκηθεί πίεση και στους άλλους φορείς για να φτιαχτεί ένας προϋπορισμός άξιος του ονόματός του. Εγώ βλέπω και ένα πρόβλημα ουσίας, το δημοσιονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Προφανώς χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις για την αντιμετώπιση του προσφυγικού η κρίση στη γεωργία, η κρίση της νεότητας και της ανεργίας των νέων. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερα κονδύλια και ούτως ή άλλως η κρίση του ελληνικού χρέους. Και όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο περικοπών. Γιατί πρέπει να χρηματοδοτηθεί και το σχέδιο Juncker, πρέπει να βρεθούν λεφτά για άλλα πράγματα. Εγώ λοιπόν διορωτώ με, μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα σκεφτούμε κάποτε ότι χρειάζεται μια νέα δημοσιονομική οργάνωση της Ευρώπης. Σωστά είπε ο Μπέγκε πριν ότι στην ουσία βρισκόμαστε μπροστά σε ε, ένα σύνολο εθνικών εγωισμών, όχι μόνο για το προσφυγικό, αλλά και για την κρίση στη Γεωργία. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ουσίας. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε πόρους, άξιους, της Ευρώπης που θέλουμε, που θέλουμε να είναι μια σημαντική δύναμη. Ίσως πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Αναμένω με ανυπομονησία να εμφανιστεί ο Μάριο Μόντι και να μας πει με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Ρώτησα και δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ. Υπάρχει λοιπόν ένα θεμοσία, όπως είπα, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εγώ θα ήθελα η Επιτροπή Προϋπολογισμών να πει καθαρά ότι έτσι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάιερ. διερωτηθήκαμε ως δημοκρατικές πολιτικές ομάδες πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και στόχος των προσπαθειών μας είναι τα όσα έχουν επιτευχθεί για την επίλυση της κρίσης των πληρωμών να μην τεθούν σε κίνδυνο. Εγώ θυμούμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι τα χρήματα που ζητήσαμε την άνοιξη θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών. Με εξέπληξε που το Συμβούλιο Υπουργών που είχε διαβεβαιώσει ότι θα το πράξει, ειδικά στην πλευρά των πληρωμών, προχώρησε σε περικοπές. Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου εδώ αλλά και σε επισκέψεις που έκανε στο γραφείο μου μου δήλωσε ότι οι περικοπές αυτές προέκυψαν από το γεγονός ότι οι αυξήσεις που είχαμε δεχτεί ήταν τόσο υψηλές ώστε δεν υπήρχε επαρκής απορροφητικότητα για να απορροφηθούν. Δεν έπεισε με το επιχείρημα αυτό. Στον κοινωνικό διάλογο στην κατηγορία 2 βλέπω ωστόσο να μειώνονται σημαντικά ποσά να περικόπτε σημαντικά ποσά που δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα απορροφικότητα. Βλέπω για παράδειγμα ο προπολογισμό του Οργανισμού για την Ισότητα των Φύλων βλέπω ότι πάνε εκεί και περικόπτουν 3.700 ευρώ. Ε, μήπως αυτό γίνεται διότι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι υπάλληλοι του Συμβουλίου των Υπουργών. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα απορροφητικότητα από πλευρά των χωρών μελών. Μόνο αν καταλήξουμε πραγματικά στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δεδομένη η απορροφητικότητα, τότε θα έχουμε και ισχύ του επιχειρήματο αυτού. Άλλωστε είπε ο Φερνάντε προηγουμένω ότι οι αυξήσει που προβλέπουμε για τον προπολογισμό ενδεχομένω θα πρέπει να μειωθούν. Κρίση λοιπόν πληρωμών. Η ερώτησή μου προ την Επιτροπή είναι εξασφαλισμένη η αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών με το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου. Αν είναι εξασφαλισμένη, τότε αυτό που είχατε πει προηγουμένως, παλαιότερα δηλαδή, ότι δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά, τότε δεν είναι, δεν είναι σωστό. Αλλιώς πρέπει να καταστήσουμε σαφές στις χώρες μέλη ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Εγώ χρειάζομαι λίγη υποστήριξη με επιχειρήματα από πλευρά τη Επιτροπής, διότι αλλιώ, θα πρέπει να πούμε στο Συμβολυπουργό ότι τα όσα είχε δηλώσει σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών, δύο μήνες μετά τα έχει λησμονήσει. Δεύτερο πρόβλημα που βλέπω είναι το ερώτημα, μάλλον πώς θα οργανώσουμε την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Μελετών. Ανάπτυξη και απασχόληση. Και τέλος, λέω τα ίδια που είπε και ο Ράιμερ Μπέγκε, τι μπορούμε, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε με τα μέσα που είναι διαθέσιμα στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των προσφύγων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζεται 6.000 ευρώ παραπάνω για κάθε πρόσφυγα, για το λεγόμενο resettlement. Αυτό σημαίνει ότι με τα νούμερα που έχουμε σήμερα για ένα μια περίοδο μάλλον ενός χρόνου και λίγο παραπάνω, χρειαζόμαστε 720 εκατομμύρια. Τώρα έχω ένα πρόβλημα συστημικό. Νομίζω το ίδιο με αυτό που είπε πριν ο Ράιμερ Μπέγκε. Ή θα φτιάξουμε έναν προπολογισμό Ανεξαρτήτως αυτού, δηλαδή θα παριστάνουμε σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα αυτό, θα προχωρήσουμε στις γνωστές ιεροτελεστικές μας ε, διαμάχες όπως κάθε χρόνο και θα πάμε βλέποντας και κάνοντας τι θα αποφασίσει το Συμβουλίο. Ή από την άλλη μεριά θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε, να προβλέψουμε κάποια κονδύλια δηλαδή που θα χρειαστούν, διότι θεωρώ ότι το Συμβούλιο Υπουργών κάποια στιγμή οφείλει να λάβει πιο ξεκάθαρες αποφάσεις και όχι να περιορίζεται στο business as usual. Διότι αν προχωρήσουμε πάλι σε εκ των υστέρων διορθωτικούς προπολογισμούς πάλι στην ουσία χάνουμε χρόνο. Θα χρειαστεί διαβούλευση του διορθωτικού προϋπολογισμού, πάλι βλέπε προθεσμίες, διαδικασίες και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο πρέπει να δράσουμε ταχύτητα. Ταχύτατα. Και επανέρχομαι στην επιχειρηματολογία του Ράιμερ Μπέγκε. Ένα πράγμα θεώρησε σωστό, σωστό. Ήρθε και με είδε ο εκπρόσωπος του UNHCR για τους Παλαιστινίους και μου είπε ότι η οργάνωση η οποία προσφέρει βοήθεια εδώ και δεκαετίες στα στατόπεδα προσφύγων τον περασμένο χρόνο μπήκε σε σοβαρότατη κρίση που ξεπεράστηκε χάρη σε χορηγήσεις των ΗΠΑ και ορισμένων αραβικών χωρών. και χρειάζεται αύξηση της δικής μας συνεισφοράς πλέον κατά περίπου 72 εκατομμύρια. Εάν δεν το πράξουμε, η οργάνωση αυτή θα μπει σε πάρα πολύ μεγάλες δυσχέρειες. Και μιλούμε εδώ για μια οργάνωση η οποία εξασφαλίζει σχολική εκπαίδευση πολλών νεαρών Παλαιστινίων. Κάτι το οποίο είναι ένα από τα τελευταία σταθεροποιητικά εργαλεία που λειτουργούν ακόμη σε αυτά τα ε, παλαιστινιακά στρατόπεδα προσφύγων. οι άνθρωποι θα σηκωθούν να φύγουν από εκεί και θα πάνε να βρουν αλλού. Αυτά δηλαδή που κάνουμε τώρα είναι πολιτική που οφείλει να προβλέψει και κάποια συμβολή στην Εγγύς Ανατολή. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα, αλλά θα πρέπει και οι αρχηγοί κατών και κυβερνήσεων να κάνουν και αυτοί, να συμβάλλουν και αυτοί. Και επειδή λοιπόν συμβαίνουν αυτά, διαρωτώ εάν και αυτή εδώ η διαδικασία του προϋπολογισμού θα ακολουθήσει την ίδια πορεία όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θα ζητούμε περισσότερα, το Συμβούλιο θα αρνείται και τελικά θα φτάσουμε Χριστούγεννα να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο θα ικανοποιεί λίγο πολύ όλου. Αυτό πρέπει να κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε συστηματικά την κρίση που, βλέπετε, που βλέπουμε να έρχεται. Δεν έχουμε τόσο χρόνο. Γιατί αν συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα, δεν λύνουμε κρίσεις, αλλά τις οξύνουμε. Ευχαριστώ. Καθένα κατανοεί την βαρύτητα τη κατάσταση. Να δώσω το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο για να μα εξηγήσει πολύ συγκεκριμένα πώ ακριβώς ε, ε, θα αξιοποιήσει αυτέ τι πιστώσει. Τι θα γίνει λοιπόν τι πιστώσει, ποιε θα είναι οι προτεραιότητες ε, για την μείωση τη μετανάστευση που να δοθούν και περισσότερα κονδύλια, για να δοθούν περισσότερα μέσα στους καταβλισμούς Τουρκία και Λίβανο. Παρακαλώ. Ο κ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ βεβαίως πρώτα τον Γενικό Εισηγητή για την εργασία που έχει καταβάλει ως τώρα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, και εγώ ωστόσο ευνηδιάζομαι λίγο από το γενικότερο περιεχόμενο και από τις πολλές ε, πτυχές που νομίζω ότι δεν δείχνουν να έχουμε εγκύψει... πραγματικά στην ουσία των προβλημάτων που εξήγησαν πολύ καλά και ο κύριος Μπέγκερ και ο κύριος Γκάιερ. Γι' αυτό να με επιτρέψετε ωστόσο να επανέλθω και να υπενθυμίσω και σε εσά κύριε Πρόεδρε και στους υπολείπους συναδέλφους ότι έχω εδώ και μήνες τονίσει ότι οφείλουμε να εγκύψουμε στο πρόβλημα αυτό. Εδώ είμαστε αναγκασμένοι να δράσουμε Πρόκειται πραγματικά για υπαρξιακό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε μέσα στη μέση μιας πραγματικής κρίσης αξιοπιστίας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατό να συνάπτουμε συμφωνίες με τις χώρες μέλη μας και αυτές κάποτε να εκπληρώνονται και κάποτε να μην εκπληρώνονται αναλόγως με τους διάφορους παράγοντες. Αφενός με την συνθήκη του Μάστριχτ φτιάξαμε ένα οικοδόμημα το οποίο δεν αξίζει πια το χαρτί που είναι γραμμένο. Δυστυχώς τώρα και με την ε, συνθήκη του Δουβλίνου ή τέλο πάντων τις συμφωνίες του Δουβλίνου έχουμε πάλι ένα εργαλείο το οποίο ίσως σαν βασική ιδέα να μην ήταν εσφαλμένο αλλά σίγουρα δεν ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες και εν πάση περιπτώσει τώρα έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκές. Ένα από τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτό ήταν ότι δεν φάνηκε αλληλέγγυα η Ευρώπη. Αυτό αναφέρεται και στη Γερμανία, την χώρα μου. Φορτώσαμε τα μεγαλύτερα βάρη στις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί δηλαδή όπου ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας για πρώτη φορά πατάει ευρωπαϊκή επικράτεια, λησμονώντας να δώσουμε τουλάχιστον κάποια αποζημίωση στις χώρες αυτές. Να μην μας εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι τότε δεν τηρούνται οι συμφωνίες του Δουβλίνου. Δεν μπορούμε ωστόσο να αρκεστούμε τώρα να πούμε «Ε, τι να κάνουμε, έτσι έγινε». Δεν αρκεί αυτό. Μου φαίνεται λοιπόν να λείπει από τούτο εδώ το σχέδιο του προπολογισμού. Μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το πραγματικά υπαρξιακό πρόβλημα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπαρξιακό πρόβλημα και για αυτού τους έρημους, τους πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια από τον προπολογισμό για τους ανθρώπους αυτού. Και βλέπω να λείπει αυτό. Χρειάζεται διάθεση πολλαπλάσιων κονδυλίων. Εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά αποτελούν ορθή επένδυση και για να διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και μια πραγματική επένδυση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οφείλει να δώσει βοήθεια, όχι όμως βοήθεια ad hoc, που ασφαλώς και απαιτείται όταν είναι απόλυτα αναγκαία. Αλλά χρειάζεται να αναπτυχθεί και ένα ευρύτερο κόνσεπτ, έτσι ώστε να μην δούμε τα κύματα αυτά να διωγγώνονται διαρκώς. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή δράση. Βλέπουμε βλέπουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες ακούγαμε να λένε στη χώρα μου, τη Γερμανία. Α, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Όσοι βλέπουν το πρόβλημα να είναι τόσο μεγάλο, στην πραγματικότητα είναι κινδυνολόγοι. Και βλέπουμε τώρα από τη μια μέρα στην άλλη να βάζουν πάλι εξωτερικούς ελέγχους στα σύνορα. Κάτι λοιπόν δεν γίνεται, κάτι, κάτι δεν πάει καλά εκεί τα ξεκάθαρα λόγια που άκουσα τώρα τα βρήκα θετικά. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίναμε ένα έγγραφο για την μετανάστευση, στο οποίο γράφουμε ότι αυτοί που ζητούν άσυλο και πρόσφυγες σε ό,τι αφορά την κατανομή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν και δικαίωμα ένστασης δηλαδή μπορούν να ενίστανται απέναντι στην κατανομή τους σε άλλες χώρες μέλη. Είναι σωστό το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε ότι σήμερα χρειαζόμαστε μία ξεκάθαρη στρατηγική, εφόσον χορηγούμε βοήθεια, η βοήθεια αυτή πρέπει να είναι και πραγματοποιήσιμη, πρέπει να είναι εφικτή. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη συζήτηση οφείλουμε να την κάνουμε εδώ στην Ευρωβουλή. Ίσως βέβαια να μην είμαστε εμείς η αρμοδιότερη επιτροπή Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αλλά οφείλουμε όλοι, όλοι να σταθούμε απέναντι στην κρίση αυτή. Και αυτά τα πράγματα εγώ δεν βλέπω να τα απηχεί ο προϋπολογισμός στο σχέδιο που λάβαμε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ διαφορετικά τα ζητήματα, είναι πολύ διαφορετικές οι κρίσεις, γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή και να ιεραρχήσουμε προτεραιότητε. Έχουμε και την κρίση των ε, προσφύγων, όμως συμφωνώ ότι πρέπει να καταργηθεί ε, και να φύγει από τη μέση το Δουβλίνο. Και μετά να δούμε και τι συμβαίνει με το κόστος. Frontex παίρνει 2 εκατομμύρια την εβδομάδα. Πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα περισσότερη διαφάνεια από αυτού. Στην Ιρλανδία, δύο άτομα από την Ιρλανδία έσωσαν, δύο σκάφη από την Ιρλανδία έσωσαν 5.000 ε, άτομα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα ποσά που δαπανώνται και αν δαπανώνται σωστά. Και πρέπει να δούμε και στις δημόσιες επενδύσεις για τις πρόσφυγες που φτάνουν εδώ και τελικά και το πολιτικό θέμα είναι πώς θα αποκλιμακώσουμε τις συγκρούσεις σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι η Συρία, και να οικοδομήσουμε μια ερευνητική διαδικασία. Και εμείς λοιπόν ως ομάδα ε, προπολογισμού πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη δική μας ιδιότητα. Και εδώ συμφωνώ ε, απολύτως με τον κύριο Φερνάντες, έκανε πολύ καλή δουλειά και η παρουσίαση του ήταν πολύ καλή και συμφωνούμε με αυτούς τους στόχους ε, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς απασχόλησης μάλιστα. συμφωνούμε λοιπόν με όλα αυτά ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Τους τελευταίου μήνε το ζητούμε με κάθε δυνατό τρόπο, γιατί θεωρούμε ότι όλες οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ε, θα απαιτήσουν αύξηση κατά ένα τρίτο του προπολογισμού, ακόμα 50 δι δηλαδή. Εκεί θα πρέπει εμεί να επικεντρωθούμε και να επιμείνουμε, να γίνει αυτή η αναθεώρηση και να βρούμε νέους και ε, επιπλέον πόρους που θα χρειαστούν και να επιμείνουμε για την ανάπτυξη της ε, δυνατότητας προχρηματοδότησης για τα κράτη-μέλη που είναι σε τόσο δυσχερή οικονομική θέση που δεν μπορούν να μπουν στη συγχρηματοδότηση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν από κοινού παράλληλα με την αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. Και βεβαίως όλα αυτά θα μας ορίσουν και ως θεσμικά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει πρώτα να θέσουμε τον άνθρωπο λοιπόν, με ανθρωπιστική προσέγγιση, με συμπόνια και αποτελεσματικότητα πρέπει να ενεργούμε. Όλα αυτά θα μας περάσουν λοιπόν στο από πού θα προέρχονται τα κονδύλια και πώ θα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, όμω νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε και κάποια στεγανά ε, για να ξέρουμε ακριβώ πού πηγαίνουμε και στην Επιτροπή εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαραγκάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ε, καταδεικνύει πολλά και σαφή. Οι επεξήγησεις του κυρίου Φερνάντες ήταν ε, πολύ θετικές και μας δείχνουν πώς πρέπει να εργαστούμε ενάντια στο ρεύμα με το Συμβούλιο και να αντιμετωπίσουμε και την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών. Η Επιτροπή αυτή έχει το έργο να επαυξήσει την Ευρώπη, να είναι η Ευρώπη επί του θέματος. Αυτό όμως δείχνει και τις αντιφάσεις ενός προϋπολογισμού που ε, θεωρείται ως ε, σύνολο των ε, μερών του και ως, όχι ως μια ευρωπαϊκή έννοια πραγμάτωσης πολιτικών με βάση τις αλλαγές που επισυμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή την οικονομική και κοινωνική κρίση ή τη μεταναστευτική κρίση που μας απασχολεί ομόφωνα. Σε λίγους μήνες περάσαμε από μία πολιτική ασφάλειας και εποπτείας που ε, συμπεριλάβανε αυτή την έννοια ε, αποδοχή στην έννοια του ασύλου. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε όχι για πρόσφυγες αλλά για πολίτες. Πολίτες με δικαιώματα που έχουν δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία και στην εργασία. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που αν θέλουμε μπορούμε να αποκρύψουμε ή να αποσιωπήσουμε. Αλλά η Επιτροπή, αυτή η Επιτροπή θα έπρεπε να προλάβει το μέλλον. Μιλάμε για καταστάσεις ε, σύραξης, είτε πρόκειται για τη Συρία είτε για το Λίβανο. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί όπως και να έχει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ολοένα και περισσότερα ε, χρήματα και με στα πλαίσια του άσυλου και της υποδοχής. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν όχι προσθέτοντας όλα ένα και περισσότερα χρήματα, αλλά επιδεικνύοντας ευελιξία μέσα στα πλαίσια του, των δημοσιονομικών αρχών, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει έναντι της εντροπίας που μας διακατήχε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, Όπω ε, όπως θα συζητήσουμε αύριο με την ε, Επίτροπο Γεωργίευα, να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 ή του συνδέοντα στην Ευρώπη, κύριε Φερνάντες. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ΚΑΠ, για το ΙΤΕΡ, που είναι μία έννοια την οποία δεν μπορούμε να αγγίξουμε πολλά ζητήματα θα ανακύψουν αυτούς τους ε, μήνες. Ελπίζω να είμαστε ε, γενναιόδοροι και ευρωπειστές. Έτσι ώστε να οικοδομήσουμε θέσεις ε, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν όλες τις ομάδες και να υπάρχει και σύνοχη όπως απαιτεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Καρδιά Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για το, τον προπολισμό 2016. Αυτό το έκανε ο κύριος ε, Γκέιερ αλλά επειδή έχουμε εδώ ενώπιον μας την Επιτροπή και επειδή μας απασχολούν οι πρόσφυγες, θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα με την Κομισιόν. Ο κύριος ε, Μαραγκάλ είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι άνθρωποι τι θα γίνει εδώ σε ένα-δύο μήνες. Δεν, είναι, δεν πρόκειται για τον προϋπολογισμό του 2016. Μιλήσαμε για ε, υποδοχή 40.000 ε, στο τέλος θα γίνουν αυτοί οι 40.000 θα γίνουν 60, 80, 120. Δείτε μόνο πόσοι φτάσαν στην Ιταλία μόνο το καλοκαίρι. Μόνο με τους αφιχθέντες ε, στην Ιταλία έχουμε φτάσει στα όρια που έχει ορίσει ο Γιούνκερ. Δεν μιλώ για αυτούς που έφτασαν στην Ελλάδα και πάνε στη ε, Μακεδονία. Μιλάμε για ένα ταμείο επίγουσας ανάγκης, αλλά δεν αρκεί. Πώς βλέπει το θέμα η Επιτροπή. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις τώρα για το τι θα κάνουμε το 2016. Εντάξει, θα μας απασχολήσει, αλλά έρχεται χειμώνας. Εάν δεν ανταποκριθούμε στην κατάσταση στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούμε, διότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση. Μιλάμε για μια καταστροφή ολκής για ένα όνειδος. Δεν χρειάζονται άλλες επεξηγήσεις ή άλλοι χαρακτηρισμοί. Θα πρέπει να μας πει η Επιτροπή πώς νομίζει ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Τι θα γίνει σε 1,5 μήνα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το Συμβούλιο να φτάσει σε μία συμφωνία. γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα ήδη. Φτάνει ο χειμώνας. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι θα συμβεί. Ο κύριος ehm, Ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία γιατί με 2.000 τροπολογίες, κύριε Ισηγητά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή σας. Τώρα, αναλύοντας τα αριθμητικά στοιχεία, αυτά που μας έδωσε ο κύριος Φερνάντες, ε, μας δείχνουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του προϋπολογισμού για να επιλύσουμε τις προτεραιότητες που ορίσαμε και νομίζω ότι ως προς τις προτεραιότητες, συμφωνούμε όλοι στις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να θίξω σε ορισμένες ε, περιπτώσεις. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις υποχρεώσεις, τις πιστώσεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξατομικεύσουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό ε, τις ανάγκες. Τα προγράμματα δηλαδή και τις γραμμές δαπάνης, δαπανών. και να προβούμε σε επιμέρους ε, μεταφορές σε κεφάλαια δαπανών που έχουν πιο επίγοντα χαρακτήρα για να επιλύσουμε τα θέματα που ανέκυψαν. Όπως είπε και ο συνάδελφος των Πρασίνων, αύριο θα έχουμε μία συνάντηση. Θα μιλήσουμε με την Επίτροπο για την απόδοση, την αποδοτικότητα του προϋπολογισμού, performance budgeting, ε, budgeting γραμμή προς γραμμή. Σε σχέση με τη μετανάστευση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι τα νέα που φτάνουν από το μέτωπο ε, δεν είναι και πολύ καλά όπως ε, απορρέουν από τη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών. Δηλαδή, μετά από τρεις μήνες από το σχέδιο Juncker, τώρα γίνεται μία επανακατανομή των 40.000 στα διάφορα κράτη. Εμείς είδαμε μόνο τα επίσημα στοιχεία φίξεων στην Ιταλία και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αρκούν τα μέτρα. Ε, καταβάλλονται ε, προσπάθειες από τους Ιταλούς φορολογούμενους για να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών μας ε, είπε ότι η διαχείριση του προβλήματος είναι πολυδάπανη δηλαδή στοιχίζει 10 ε, δις ευρώ, αν μπορούμε να ποσοστοποιήσουμε, που επιβαρύνει τους δικούς μας ε, φορολογούμενους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει κάτω από 10% σε αυτό το αριθμητικό στοιχείο και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Βεβαίω είμαι ο πρώτος που λέω ότι με 150 δις δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα της Ευρώπης, αλλά ας δούμε τα προγράμματα ή τους, ε, τις πιστώσεις που δεν έχουν απορροφηθεί και ας γίνει σωστότερη χρήση τους. Νομίζω ότι η αναθεώρηση του πολιετούς αποτελεί μία ευκαιρία για να δούμε πολλά πράγματα. Γιατί είναι απολύτως αναγκαία, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα και εμείς και οι ε, Κομισιόν αλλά και το Συμβουλίο και τα κράτη-μέλη ίσως θα πρέπει να έχουν πιο σαφείς ιδέες. Γιατί αν δούμε τις προτάσεις του Συμβουλίου βλέπουμε ότι υπάρχουν γραμμές του προϋπολογισμού που γίνονται μεγάλες περικοπές και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Άρα βλέπω ότι δεν υπάρχει θέληση από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν αυτά τα σχέδια. Και επ' θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε την όλη μας προσέγγιση, να έχουμε πιο συνεκτικές πολιτικές και αλληλένδετες με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ε, συνεκτικός με το έργο μας ή το ενδυνάμει έργο μας. Σήμερα και μπροστά σε αυτή την κρίση Μπορούμε εμείς να δίνουμε 5 δις ε, για 7 χρόνια στην Τουρκία, η οποία, ε, η οποία να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε ζητήματα όπως η μετανάστευση. Ξέρω ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνο η Επίτροπη Προϋπολογισμών, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της Επίτροπής μας και των κρατών μελών και της Κομισιόν για τον ορισμό των πολιτικών. Επίσης έχουμε κεφάλαια δαπανών που είναι πολύ σημαντικά για βοήθεια προς τον τρίτο κόσμο. Ωραία, να βοηθήσουμε τον τρίτο κόσμο γιατί είναι σε χειρότερη θέση από εμάς, αλλά πολλές φορές αποστέλουμε χρήματα για να βοηθήσουμε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της δράσης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν καλύτερο συντονισμός έτσι ώστε αυτοί οι πόροι να αποστέλλονται όχι μόνο σε αυτές τις χώρες. Η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική για να μην δημιουργεί ίδια κρίσεις ή καταστάσεις ε, φτώχειας και να επιλύονται καλύτερα προβλήματα όπως οι μεταναστευτικές ροές και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ε, άλλοι ομιλητέ. Νομίζω, κύριε Γενική Συγητά, ότι και οι προτεραιότητέ σα γενικά εγκρίνονται και από του υπόλοιπου ε, συναδέλφου. Ε, αποτελούν αντικείμενο συνένεση, όμω όλοι αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση. Και δεν μπορούμε να προδικάσουμε όλες τις επιπτώσεις και πραγματικά επικρατεί μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε και τα μέσα που θα αξιοποιήσουμε από αύριο. Πώς μπορούμε με ένα 7 ετέ, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πλαίσιο που εντάξει έχει κάποια συνέχεια, όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κρίση ανευπροηγουμένου. Και έχουμε τη δυνατότητα, την εντύπωση, προσπαθούμε να το λύσουμε με πολύ περιορισμένα μέσα. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να πάρει το λόγο, γιατί της ετέθησαν πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που ετέθησαν. Επιτρέψτε μου να μιλήσω αγγλικά. Ο κύριε Βέγκε ρώτησε κατά πόσο τα στοιχεία ε, μεταξύ των πακέτων Μαΐου και Ιουνίου συνάδουν μεταξύ τους. Ισχύει, γιατί για τις 40.000 μετακαταστάσεις του Μαΐου ο αριθμός αυτός που αποφασίστηκε ήταν 240 εκατομμύρια. Τώρα στο νέο πακέτο 120.000 μετακαταστάσεων, το ποσό είναι 720, τριπλάσια δηλαδή του προηγούμενου, συν το κόστος της ε, μεταφοράς, το οποίο δεν είναι συμπεριλαμβανόταν στο προηγούμενο πακέτο. Να επισημάνω ότι δεν είναι τα, τα μοναδικά στοιχεία του προπολογισμού. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο της μετεγκατάστασης. Δεν υπήρχε αυτό προηγουμένως. Ούτε στο πνεύμα, ούτε στο γράμμα Τη προσέγγιση του Δουβλίνου υπήρχε κάτι τέτοιο. Στο προπολογισμό έχουμε δύο κονδύλια. Έχουμε το Ταμείο ε, Ασύλου, μετανάστευση και ε, ένταξη και μετά έχουμε και το Ταμείο Εστερικής ασφάλεια. Και τα δύο από κοινού ανέρχονται σε πάνω από ένα δι, το οποίο κατανέμεται στα κράτη-μέλη. Κάθε κράτο μέλος λοιπόν πρέπει να παραδώσει επιχειρησιακά προγράμματα για να ανταποκριθεί στην ε, πρόκληση της κοινή διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι μια κοινή δράση που θα πρέπει να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί ε, στη βάση, σε συνδυασμό με τα κράτη-μέλη. Είναι αυτά τα τρία προγράμματα μαζί με τα προσωρινά μέτρα μεταγκατάσταση που έχουν προταθεί. Κατά κάποιον τρόπο έτσι θα μας βοηθήσει αυτό να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Τώρα, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος ο στην Ολομέλεια, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, υπάρχει και αυτό το Trust Fund, το καταπίστευμα για την ε, Αφρική, συμπεριλαμβανομένη και της Βορείου Αφρικής, το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί με πιο στοχευμένο τρόπο σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τρίτε χώρε, είτε είναι χώρε προέλευση είτε διαμετακόμιση, διέλευση μάλλον των μεταναστών. Θέλουμε να εισαγάγουμε ένα στοιχείο ενισχυμένη συνεργασία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Με αυτό απαντώ σε κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε, για παράδειγμα, ο κύριος Ζάνη στην παρέμβασή του. κύριος Γκάια ρώτησε κατά πόσο οι περικοπές στις πληρωμές ε, αντιστοιχούν με ε, το σχεδιασμό περιπληρωμών και τη σταδιακή κατάργηση. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιοποιήσει όλα τα επιχειρήματα και παραδείγματα για να καταδείξει ακριβώ αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αιτιολογούνται από την δυνατότητα απορρόφησης. Αν δείτε ε, τα στοιχεία της εκτέλεσης. Δεν ε, τεκμηριώνεται αυτό από πλευρά στοιχεία και νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να αποδείξουμε ότι οι ανάγκες αυτές ευσταθούν και μπορούμε να τις τεκμηριώσουμε και θεωρούμε ότι υπάρχουν τα κατάλληλα επιχειρήματα. Αυτά ήταν τα κύρια στοιχεία που σημείωσα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν έχω παραλείψει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Φαζά. Χωσέ Μανουέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για όλες τις ε, παρεμβάσεις. Ε, νομίζω ότι συμβαδίζουμε. Δεν έχουμε το Συμβούλιο μαζί μας, ε, εδώ τον μεγάλο έλεγχο γιατί η Επιτροπή έδρασε, το Κοινοβούλιο επίσης και το Συμβούλιο είναι ουραγός. Το Συμβούλιο θα πρέπει να προβάλλει μια κοινή πολιτική σε αυτή την ροή των μετανοστών. Θα έπρεπε να έχει ενωτική στάση, αλλά υπάρχει ε, μεγάλη αναισθησία μπορώ να πω και διαφορά απόψεων, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Πώς μπορεί το Συμβούλιο να έχει μειώσει μέσα τα οποία σχετίζονται άμεσα με, αυτή το, αυτό το θέμα της κρίσης, της μεταναστευτικής ε, κρίσης και των ροών. Το Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να δείξει κατά πόσο θέλει να κάνει μια επιπρόσθετη προσπάθεια, γιατί μιλάμε για μια κατεπίγουσα κατάσταση. Χρειάζονται επιπρόσθετη πόροι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Όταν μιλάμε για το κεφάλαιο 3 και το 4, μιλάμε για πολύ μικρά κεφάλαια, για πολύ μικρούς τομείς. Μιλάμε για 150 δις ενώ η 4 στις υποχρεώσεις έχει 2.690. Στα 150 δις, μα σοβαρολογείται. Δηλαδή έκοψε 8 εκατομμύρια από τα 8 δις από τα 150. Μα σοβαρολογούμε τώρα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι ε, κάνει το Συμβούλιο. Δεν καταβάλει καμία προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε μία έκτακτη κατάσταση. Δεν θα μπω στη λογική της κοινή ε, πολιτικής και του κοινού μετόπου που είναι προαπαιτούμενο. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Δηλαδή το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία δυστυχώς θα είναι πρόσφορο έδαφος για τους ε, τρομοκράτες, εάν δεν επιλύσουμε αυτό το θέμα, για να προχωρήσουμε. αλλά θα ήθελα να μιλήσω τώρα συνολικά για το σχέδιο προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας ε, λόγια. Οι δικές σας ανησυχίες είναι και δικές μου ανησυχίες και αντικατοπτρίζονται στις ε, προτάσεις που έγιναν, ιδιαίτερα στις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Και με γνώμονα αυτή τη φιλοδοξία θα προχωρήσουμε σε μια ευρύτερη συνένεση εδώ στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα επιδείξει διαφορετική στάση. Έχω βρεθεί σε πολλές ε, ε, συναντήσεις συνδιαλλαγής όπου το Συμβούλιο έδειξε μία ευαισθησία πολλές φορές. Ενώ άλλες φορές δεν ήθελε να δράσει καθόλου. Ήθελε να αναβάλει το θέμα και να προβάλλει μεσοβέζικες λύσεις. Πολλές φορές το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν υφίσταται το πρόβλημά μας και αυτό το είπατε και εσείς. Φτάνει πια με αυτή τη στάση του Συμβουλίου. Ελπίζουμε αυτή η φωτογραφία του παιδιού στις ακτές της ε, Τουρκίας να μην διαγραφεί από τη συλλογική μας ε, μνήμη. Θα πρέπει να δράσουν η αρχηγοί κρατών επί της ουσίας, έτσι ώστε οι αξίες μας, οι αξίες της αλληλεγγύης και της ευθύνης να ισχύσουν ε, έμπρακτα. Η αλληλεγγύη φαίνεται έμπρακτα, μέσω δράσεων. Δεν ε, μπορεί να είναι μόνο δηλωτική και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Βεβαίως δεν θα αλλάξουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά οι τροπολογίες των συναδέλφων, των συναδέλφων καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής του πολιετούς. Θα πρέπει να έχουμε πιο ευέλικτα μέσα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην κρίση που μας απασχολεί. Αυτό είναι, αυτή είναι μια νέα φάση. Ας επικεντρωθούμε στον προϋπολογισμό το 1% του, ε, των εθνικών ΑΕΠ και ας ελπίσουμε να επιβιώσει η ελπίδα και η φλόγα της ελπίδας να μην σβήσει. Merci, Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε μια σαφή θέση μαζί με το Συμβούλιο, με σαφείς προτεραιότητες. Για να είμαστε πιστικοί απέναντι στο Συμβούλιο πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο ενωμένοι και κάπως να συγκεράσουμε αυτές τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων που βεβαίως συνιστούν και τον πλούτο της Επιτροπής μας αναφέρθηκε πολύ το θέμα της ε, συνοχής. Άκουσα ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, στοχεύσει καλύτερα την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά για να γίνει αυτό από τις χώρες που υποφελούνται αυτής της βοήθειας μπορούμε να λάβουμε τη δέσμευση ότι θα περιορίσουν ε, τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη σε αντιστάθμισμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Και Εάν αυτή η χώρα δεχθεί ότι οι πίκοοι της χώρας αυτής, οι οποίοι ξαφνικά θα βρεθούν στην Ευρώπη, θα επιστρέφονται απευθείας ε, στη χώρα. Υπάρχει αυτή η συνέπεια. Ναι, Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η πρόθεσή μας υπάρχει ένα στοιχείο συντονισμού και συνεργασίας στα προγράμματα ανταξιακής βοήθειας ε, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις, ε, τη συνεργασία στα σχέδια για την επιστροφή ή για την ε, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Για να έχουμε λοιπόν ένα πιο έντονο τέτοιο στοιχείο στις συμφωνίες που θα συνάπτουμε με αυτές τις χώρες. Επομένω, θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση, αξιοποιώντα υφιστάμενα μέσα, αλλά τα οποία θα ε, ομαδοποιούνται και θα ταξινομούνται με πιο ξεκάθαρο τρόπο για να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε τις μετραστικές ροές. Προσπαθούμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα στοιχεία και αυτό να μας ε, να επιτρέψει και τη χρηματοδότηση ταχύτερη χρηματοδότηση και σύσταση ε, τέτοιων ε, δράσεων, να έχουμε και εμείς μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να κλείσουμε και αυτή τη συζήτηση για τον ε, προπολογισμό του 2016. Θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα Θα δούμε λοιπόν ε, τη θέση μας απέναντι σε αυτές τις τροπολογίες. Επανερχόμαστε στο 2015 και τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρδιά Ζάπαλ. Ευχαριστώ. Ε, ένα μόνο λεπτό για να σας πω γιατί ε, μιλάμε με αυτό το διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 6. Υπάρχουν υπάρχουν ε, νέες, ε, νέες εισφορές, ε, ιδιαίτερα στον τομέα της ζάχαρης και τελωνιακά έσοδα. Μιλάμε για υψηλότερα πόσα σε σχέση με το 2014. Γι' αυτό χρειάζεται, δεν χρειάζεται να ζητήσουμε τόσα πολλά χρήματα από τα κράτη-μέλη ως προς την εισφορά τους δεν χρειάζεται να αποδώσουν ε, τα 2.260.000 ευρώ. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτή η επιστροφή με βάση τα νέα έσοδα. Επίσης, η Επιτροπή μας προτείνει δύο νέες γραμμές στο, στην αναπτυξιακή πολιτική που δεν έχουν ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Απλώς για... υπάρχουν αυτές οι δύο νέες γραμμές ως προς το καταπιστευματικό ταμείο και δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν διορθωτικό προϋπολογισμό με δύο μικρές ε, τεχνικής υφής ε, τροποποίησεις που δεν έχουν καμία επίπτωση Προτείνω λοιπόν να εγκρίνεται χωρίς ε, τροπολογίες αυτές τις διορθώσεις που θα εγκρίνει και το Συμβούλιο με τη σειρά του, χωρίς προβλήματα πόσο γνωρίζω. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Ακολουθούμε λοιπόν ε, την πρόταση της κυρίας Γκαρδιά Ζάμπαλα. Οι τροπολογίες για το προσχέδιο προπολογισμού θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι και θα τις εξετάσουμε στην Επιτροπή μας εδώ τις 12-13 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια θα περάσουν 26 έως 29 Οκτωβρίου. Κύριε Μαργάλη, παρακαλώ. Όχι, στα επόμενο σημείο. Ξανά με κύριες Μπάνα. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο για την ε, κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην ε, Παγκοσμιοποίηση. Ε, μια υπόθεση που αφορά την Αλιτάλια και ο κύριος Μαραγκάλ αντικαθίσταται την κυρία Μόνικα Βάνα. Εντάχει, εξ ονόματος κυρίας Βάνα που δεν είναι παρούσα σήμερα, πρόκειται για μια διεκπαιρέωση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στη παγκοσμιοποίηση για μια αίτηση της Ιταλίας ε, και που αφορά την Αλιτάλια. Πρόκειται για ένα θέμα ίσονο σημασίας σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων. Πρόκειται για 2,3 εκατομμύρια ευρώ Άρα η συνεισφορά είναι της τάξης του 1,4 εκατομμυρία. Μιλάμε για 154 εργαζόμενους για να μπουν στην αγορά εργασίας. Αρχικά ήταν 1249 οι εργαζόμενοι, γι' αυτό μιλάμε και για μια πολύ μικρή ποσοστή αναλογία. Ε, ξέρετε για την κατάσταση της ε, Αλιτάλια. Δυστυχώς συρρυκνούται η δράση της, ιδιαίτερα μετά το 2008. Η αίτηση της ε, Ιταλίας τηρεί τα προαπαιτούμενα και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε αυτό το αίτημα της Ιταλίας, δηλαδή να ισχύσει, να τεθεί σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ε, λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση. Ε, ευχαριστώ. Έχω κάποια εμπειρία από σχετικές υποθέσεις στο παρελθόν. Θυμούμε την υπόθεση Μαρή Ντικρό αρχών του έτους. 0,3% είχαν διοικητικές δαπάνες για την χορήγηση αυτής της βοήθειας. Ενώ στην περίπτωση της Αντιτάλια, βλέπω 4% διοικητικό κόστος του συνολικού ποσού που θα εκχωρηθεί από το Ταμείο Προσαρμογής στην Κινητικότητα. Βλέπω λοιπόν ότι είναι 13 φορές ακριβότερο από το άλλο. Ε, έχω την περιέργεια γιατί. Ξαναλέω, η υπόθεση Μαρίτικρό 0,3% ε, του, του συνόλου του ποσού. Για την Αλιτάλια βλέπω, όπως είπα, το 4% ε, που είναι 13 φορές περισσότερο. Κύριε Μαντραγκάρ. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες της υποθέσεως αλλά μάλλον οφείλεται στο μικρό συνολικό ποσό. Το διοικητικό κόστος ε, συνήθως είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Εμένα δεν με εκπλήσει. Μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο σε ποσοστό, αλλά το συνολικό ποσό δεν είναι σημαντικό. Εμένα μου φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Μήπως, λέει ο Πρόεδρος, μπορεί ε, να συμβάλλει στην διευκρίνηση του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το 4% είναι ε, ένα ενδεικτικό επίπεδο ποσού το οποίο προτείνει ε, γενικώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα αν η χώρα μέλος μπορεί να δώσει άλλη πρόβλεψη αυτό απαιτεί να μπορεί να ανοιχνευτεί ο τρόπος ανάλυσης του ποσού αυτού και να δικαιολογείται η δαπάνη του. Σε άλλες σχετικές υποθέσεις οι χώρες μέλη δεν μπόρεσαν να αιτιολογήσουν αυτό το διοικητικό κόστος και επομένως το ποσοστό της διοικητικής δαπάνης κρατήθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο από το ποσοστό που ζητούσε η χώρα μέλος. Μάλιστα, αυτό αποτελεί αρχή απαντήσεω, κύριε εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Η κυρία Γκρέσλε, μην ανησυχείτε, θα τα εξετάσει όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένη να ομιλεί με τον Γενικό Εισηγητή. Άλλο κανεί δεν ζητεί το λόγο. Κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, εξέταση και ψηφοφορία επί των τροπολογιών στην περίοδο συνεδριάσεως 28-30 Σεπτεμβρίου. Είπα 28 πάλι. Όχι, 23 είναι η προθεσμία προφανώς για την κατάθεση. Alors, με την Ελλάδα και με τα όσα βρέθηκαν στον πυρήνα της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των ελληνικών αρχών. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, δηλαδή επ' αυτών έχω υποβάλει σχέδιο επιστολής που έχετε λάβει γνώση που περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Προπολογισμών. Έχετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής. Μπορώ να θεωρήσω ότι την εγκρίνεται, εγκρίνεται από πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Προπολογισμών. Εσείς κύριε Κέρμελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου φαίνεται Ορθή η επιστολή σας, απηχεί τα όσα συζητήσαμε, ωστόσο σε ένα σημείο της οφείλω να ομολογήσω ότι θα επιθυμούσα να επέλθει μία διόρθωση διότι υποβάλλουμε αληθινά ερωτήματα στην επιστολή κάνουμε όμως την εισαγωγή στα ερωτήματα αυτά με την διαπίστωση ότι κάνουμε τις χορηγήσεις αυτές χωρίς προϋποθέσεις. Όταν ωστόσο υποβάλλουμε τα ερωτήματα αυτά, πρέπει αυτά να έχουν και κάποιες συνέπειες. Δηλαδή να διατυπώσουμε τις ερωτήσεις αυτές λέγοντας ότι θα συμφωνήσουμε με τις ε, παροχές εκ μέρους μας εφόσον ικανοποιηθούν τα ερωτήματά μας, εφόσον δηλαδή απαντηθούν ικανοποιητικά οι ερωτήσεις μας αυτές. Ο πρόεδρος δεν έχει μικρόφωνο ανοιχτό. Ως τώρα δεν έχω βρει εναλλακτική διατύπωση. Ποια είναι η συγκεκριμένη πρότασή σας για το σημείο αυτό της επιστολής. Ähm, ο κύριος Κέρμερ, ε, ε, ο πρόεδρος, όχι, ο κύριος Κέρμερ. Ευνηδιάζομαι τώρα, δεν έχω ε, σχέδιο διατυπώσεως, Ευχαριστώ αν θέλετε. Αλλά αν θέλετε να εξοικονομήσουμε χρόνο, αυτό που θα προτείνω είναι να το συζητήσουμε. Εγώ δηλαδή θα ήθελα η έγκρισή μας να εξαρτηθεί από την ικανοποιητική απάντηση των ερωτήσεων μας. Αυτό δηλαδή με απασχολεί βασικά. Επαναλαμβάνω, η παρατήρησή σας αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων στην προκατακτική φάση διατυπώσεως του κειμένου και τελικώς όμως ε, δεν υποστηρίχθηκε από πλειοψηφία. Κύριε Φερνάντες, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με την βοήθεια προς την Ελλάδα. Εν τέλει πρόκειται για μια επιστολή ε, συμβατική. Εάν δηλαδή συμφωνεί με τις προβλέψεις των κανονισμών ή όχι. Και για να δοθούν τα χρήματα αυτά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και αυτές δεν μπαίνουν στην επιστολή. Προχωρήσαμε και λίγο περισσότερο με ερωτήσεις που δεν συνδέονται απολύτως με το θέμα. Κατανοώ λοιπόν την θέση του συναδέλφου μας. Νομίζω όμως ότι η επιστολή είναι έντονα διατυπωμένη, δείχνει και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό. Πρέπει ωστόσο να δούμε ένα πράγμα. Είναι ουδέτερο το περιεχόμενο. Μάλλον δεν πρόκειται για νέο χρήμα. Μπαίνει, εντάσσεται μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή γίνονται σεβαστοί οι κανόνες η θέση και η επιστολή του Προέδρου είναι επαρκώς ισχυρή για να δείξει ότι ποιες είναι δηλαδή πραγματικά οι ανησυχίες της Επιτροπής Προεπολογισμών. Κοιτάξτε, όλα θα αποτελέσουν θέμα ελέγχου τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Και ίσως θα χρειαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάει και να δει επιτόπου τι γίνεται στην Ελλάδα, χωρίς να περιμένει την παρέλευση προθεσμιών. Είναι υπόθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά είναι και υπόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πάει να δει τι γίνεται. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να τα πει και δημοσίω. Δεν είναι μονάχα υπόθεση τη Τρόικα ή των θεσμών. Τώρα νομίζω ότι η δυσχέρεια θα εντοπιστεί στην πραγματική υλοποίηση των δεσμεύσεων. Αν κυριε συγχωρείτε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημειώνω πρώτον ότι την επιστολή δεν την βρίσκω στους φακέλους μας. Το βρίσκω λυπηρό αυτό, διότι είχε συμφωνηθεί ότι θα περιληφθεί στα ντοσιέ μας και το βρίσκω σημαντικό. Μόλις τώρα βλέπω την επιστολή. Θα ήθελα να μπορούσα να την είχα μελετήσει περισσότερα και προσεκτικότερα. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θα μεταβεί στην Ελλάδα από τις ε, 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα. Θα δούμε 5 από τα 181 έργα και που δεν πετύχε να ολοκληρωθούν μέσα στην πενταετία. Όσο μεγαλύτερα είναι τα έργα, τόσο μεγαλύτερη και η αποτυχία. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά μην θεωρήσετε ότι τα πολλά χρήματα βοηθούν και πολλά. Εγώ θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τούτο εδώ το πακέτο βοήθειας να το διατυπώσει έτσι πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή 100% χρηματοδότηση για τα χρήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνοι. Αλλά ό,τι πάει στο κράτος, εκεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Διότι αυτό εξαρτάται από το πόσο υλοποιήσιμο είναι το έργο και έχω πάρα πολλές αμφιβολίες και ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης ορισμένων έργων. Και δεν εξυπηρετούμε ούτε το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε εν τέλει και της Ελλάδας, εάν δεν το προσέξουμε αυτό. Εν ώψη των βασικών αυτών προκλήσεων και της διοικητικής ικανότητας, όπου έχει πάρα πολλά κενά και τελικά από αυτούς θα εξαρτηθεί η σωστή απορρόφηση των χρημάτων. Νομίζω ότι ολόκληρο το πρόγραμμα δεν ικανοποιεί του στόχου του. σω μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει λίγα λόγια ακόμα. Δηλαδή ποιο θα στηρίξει την ελληνική διοίκηση εφόσον δεν επιτρέπεται να συνεχίσει το έργο τη η Task Force. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνεται κάποια συμβιλική διατύπωση ότι υπάρχει λέει μια high level group. Ποιο όμω θα ενισχύσει την ελληνική διοίκηση για να υλοποιήσει τα έργα αυτά δίνονται παραπάνω λεφτά στην Ελλάδα και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι οι άλλες χώρες λαμβάνουν λιγότερα. Γιατί κάπου θα λείψουν αυτά τα πράγματα. Εγώ βλέπω τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι δεν έχει θεματοποίηση και αυτές τις επιπτώσεις στους υπολείπους. Και μιλώ και για τις πιστώσεις και για τις υποχρώσεις. Εν τέλει συμφωνώ ότι είμαι ικανοποιημένη δηλαδή ότι εδώ περιορίζεται μονάχα στην Ελλάδα, αλλά ξαναλέω ότι εάν δεν δοθεί συγκεκριμένη βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εν τέλει αυτές θα φροντίσουν για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Για την επιστολή, ο πρόεδρος. Σας έχει έρθει κανονικά στη γραμματεία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την προηγούμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω ότι η γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών διαβίβασε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών την επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι όμως στους φακέλους κύριε Πρόεδρε. Σας διαβιβάστε. Πρόκειται για επιτάχυνση πληρωμών χωρίς όμως να εμπλέκονται πρόσθετα κονδύλια. Δηλαδή δεν αφαιρούνται κονδύλια από άλλες ε, από άλλα πράγματα. Τώρα, επί της ουσίας δεν θα με εκπλήξει να επανέλθουμε σε έξι μήνες, διότι όταν αναλαμβάνεται μια δημοσίευση, ε, αναλαμβάνεται μια δέσμευση μάλλον, της τάξης του 3% πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2016, αυτά τα πράγματα ούτε στα θαύματα δεν γίνονται. Μπορεί σιγά σιγά να εξαφανιστεί αυτή η παράλληλη οικονομία στην Ελλάδα. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες συναδέλφους μας έτσι ώστε να φροντίσουν και αυτοί να αλλάξουν οι συμπεριφορές αλλά δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι δύσκολο και θα χρειαστεί διαρκής έλεγχος αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένοχη διότι, και ιδίω η Ευρωζώνη, διότι άφησε απολύτω να κάνει ο καθένα ό,τι ήθελε επί μια δεκαετία. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, διότι δεν φρόντισαν να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Όλε οι χώρε. Κανένα έλεγχο, καμία α, τήρηση των δεσμεύσεων. Και οι βασικοί πιστωτέ τη Ελλάδα είναι πάλι Ευρωπαίοι. Και όταν δίνετε πίστοση σε κάποιον, είστε και εσεί υπεύθυνο. Ο καθένας λοιπόν έχει τις ευθύνες του στην υπόθεση αυτή και κάπως πρέπει να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, φροντίστε να είναι οι κάρτες σας στην ε, σχισμή. Θα κάνουμε πρώτα μια ε, δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε ότι όλα λειτουργούν καλά, αρχίζει. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται ακόμα για την πραγματική επίσημη ψηφοφορία, μόνο θέλουμε να δούμε αν λειτουργούν καλά οι συσκευέ σα. Κυρία Χόλμπαϊερ, δεν λειτουργεί το, το μηχάνημα. Μάλιστα. Έχει αρχίσει λοιπόν η διαδικασία της ψηφοφορίας. Επανέρχομαι στην αφιτηρία και ρωτώ Όσοι εγκρίνουν την επιστολή, παρακαλώ να ψηφίσουν υπέρ. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Τέλος. ...22 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Ακολουθεί το επόμενο. κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για καταστροφές στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα το 2015. Εδώ δεν υπάρχουν τροπολογίες. Θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. 25 ψηφίσατε, 24 υπέρ και μία ψήφος κατά. Τμήμα 3 του προπολισμού 2015, κυρία Γουάρδια Ζαβάλ. Έχουμε τρεις μεταφορές. Η πρώτη είναι 26, όπου ζητάμε 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πλαίσια των ε, πληρωμών ε, ως προς βασικές ανάγκες, ανάγκες στο τομέα υγείας και υγιεινής ε, νερού και λοιπά στο νότιο Σουδάν. 27 που είναι 20 εκατομμύρια υποχρεώσεις και 19 στις δαπάνες πληρωμών για να βοηθήσουμε την Ούναρα, την Παλαιστινιακή Αρχή τους Παλαιστίνιους για να πληρωθούν 22.000 ε, καθηγητές και οι 28 για 42 εκατομμύρια ευρώ, 10.000 για τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στη Συρία, 20 για τους Σύριους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λίβανο και στην Ιορδανία, 10.000 ε, για ανθρωπιστική βοήθεια για τη Συρία και 5 για το Ιράκ. Γι' αυτό μιλάμε για 45 εκατομμύρια ευρώ. Ζητώ την συνένεσή σας ε, επιγόντως. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις, ε, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ψηφίζουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε και τις τρεις μεταφορές. Έχετε αντίρρηση. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία για τις τρεις μεταφορές. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, μία ψήφος κατά, εγκρίνονται οι πιστώσεις, άλλα τμήματα για το 2015 Χολμάιερ. Έχετε προτάσεις μεταφοράς για το ελεγκτικό. ΕΟΚΕ και ΕΙΕΒ. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, δίκιο έχετε. Και πρώτα το ελεγκτικό συνέδριο. Μιλούμε για μεταφορά πιστώσεως 690.000 ευρώ. από τον τομέα των ε, μισθών και αποζημιώσεων, διότι ορισμένες προσλήψεις έγιναν στο τελευταίο τρίμηνο του 2015 και επομένως περισσεύουν κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα τα χρειάζομαστε τώρα αφενός για εξοικονόμηση κόστους ενέργειας, περίπου 160.000 ευρώ. Δεύτερο πόστο, συντήρηση. Στην περίπτωση αυτή για τον κλιματισμό ορισμένων τμήματων του κτηρίου του ελεγκτικού συνεδρίου στον χώρο συσκέψεων και στο κτίριο K2. Τρίτο, πρόκειται για την προσαρμογή των συστημάτων πληροφορικής ε, για ένα κόστος 170.000 ευρώ, σύνολο 690. Το άλλο είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Μιλώ για μια μικρή μεταφορά 40.800 ευρώ από τον ε, τομέα εξωτερικής ανάθεσης μεταφράσεων για να μεταφερθεί σε ε, συντήρηση συστημάτων ηλεκτρονικής μεταφράσεως και ορισμένων γραφείων. Ο τρίτος τομέας αναφέρεται στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Πρόκειται για 3.763.000 ευρώ που θα αφαιρεθούν από έξοδα μισθώσεων, για μισθώσεις δηλαδή, διότι έγιναν και προσαρμογές των μισθών από το 2012 έως 2014 και εκεί υπάρχουν ορισμένα, ορισμένες ε, συγγνώμη, ορισμένα πλεονάσματα που θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την αντιμετώπιση του κόστους που έχει προκύψει από το χαμηλότερο ευρώ. Χαμηλότερο ευρώ σημαίνει λόγω μεγαλύτερης διαφοράς από το αμερικανικό δολάριο προβλήματα στην ε, μισθοδότηση ορισμένων ε, μελών του προσωπικού της υπηρεσίας σε άλλες χώρες. Πρόκειται για 1.800.000. Ένα άλλο ποσό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Paymaster ανέλαβε και άλλες δαπανές αφενός για, το, για την πληρωμή του λογισμικού για την διοίκηση του προσωπικού και τρίτο, διαχειρίζεται τώρα τα οικονομικά περισσότερων μελών του προσωπικού. Τέλος, 200.000 για οικογενειακά επιδόματα, οικογενειακές παροχές, που είναι υψηλότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Και τέλος, 10.000 ευρώ για μια υποτροφία ενέδωσης ε, πρακτικής άσκησης ενός πτυχιούχου και τέλος για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, εγώ ξαναμίλησα σήμερα με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων σήμερα το πρωί, για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου για την ύπατη εκπρόσωπο για ζήτημα της Κολομβίας, για ζήτημα της Κολομβίας, διότι συζητούνται αυτή τη στιγμή ζητήματα προξενικών θεωρήσεων με την χώρα αυτή και επομένως για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονος. Τώρα κάτι άλλο το οποίο ε, ναι μεν λέμε ότι ε, οι χώρες μέλη ζητούν περικοπές, κάνουν τις περικοπές αυτές όμως ε, στις συμβολές τους στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων για παράδειγμα για αποσπασμένους στρατιωτικούς ε, συμβούλους αρχίσαν από την ε, ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων, τώρα προχωρούν σε περικοπές στις ε, παροχές τους στο, προσωπικό, στο στρατιωτικό προσωπικό που αποσπούν. Εκεί πρόκειται για 200.000 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. 400.000 ευρώ προχωρούν σε μέτρα ασφάλειας 95.000 καθίστανται αναγκαίες λόγω της καταστάσεως ασφαλείας και της στρατιωτικής καταστάσεως διότι αυτές καθιστούν αναγκαίες νέες δραστηριότητες από την ύπατη εκπρόσωπο και τέλος 216.000 είναι νομικές δαπάνες και αποζημιώσεις διότι το αρχικό ποσό των 25.000 που είχε προβλεφθεί φάνηκε πάρα πολύ μικρό. Εν τέλει λοιπόν 3.763.000 το σύνολο του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Οι παρατηρήσει σας για την ε, εξωτερική δράση πράγματι χρειάζονται μέσα. Αλλά πώς ε, γίνεται αν υπάρχει ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Όχι αρκετή, λέει η κυρία Χολμάιερ. Καθόλου θα έλεγα εγώ. Υπάρχει εξωτερική παρουσία. Έχουμε 28 και ακόμα μία, μια 29η. Ναι, και πραγματικά πρέπει να γίνουν εξοικονομήσεις. 3.000 συνεργάτε νομίζω για την εξωτερική δράση, Χωρί να υπάρχει εξωτερική πολιτική. Έχουμε μια ευρωζώνη που κανονικά να υπάρχει μια πολιτική του ευρώ, αλλά δεν υπάρχει καν ε, αντίστοιχο Υπουργείο, με το οποίο θεωρώ παράδοξο. Και εδώ κλείνει η παρένθεση. Α ε, ψηφίσουμε τις πιστώσει για κάθε θεσμικό όργανο, συμφωνείτε και εσεί αρχικά για το ελεγκτικό συνέδριο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ, μία κατά, δύο εποχές Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Κυρία Χολμέιερ, για τα ακίνητα, φαντάζομαι δεν υπάρχουν αιτήματα. Επιβεβαιώνει η κυρία Χολμάιερ. Επομένω, φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή τη διάταξη. Ραντεβού αύριο στι 9 το πρωί για να συνεχίσουμε τι εργασίε μα. Θα έχουμε κοινή ακρόαση Επιτροπή Προπολογισμών και Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η ελέγχου του προπολογισμού, μάλλον. Και θα σε προεδρεύσει και η κυρία Γκρέσλε μαζί με μένα. Είστε πανεδίνοι.